Dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλούμε ε, να ξεκινήσουμε την εκτή μας συνεδρίαση. To the Yuri colleagues, as... Ε, Καλώς ήρθατε συνάδελφοι από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Όπως τα γνωρίζετε, Θα έχουμε την πρώτη εξέταση της έκθεσης ενός πολύ σημαντικού θέματος και πολύ αναμενόμενου. Μεγαλύτερη φορολογική διαφάνεια και δημόσιος έλεγχος των εταιρικών φόρων. Μεγάλη μα χαρά που μπορούμε να συνεργαζόμαστε με του συναδέλφου τη Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων βάσει του άρθρου 55 του εθνικού Κανονισμού για το θέμα αυτό. Και είμαστε πολύ σαφείς ως προ το θέμα τη νομική βάση αυτή τη νομική πρότασης. Έχει να πει κάτι, Μαντλέν. Νομίζω ότι έχουμε λίγο χρόνο να ξεκινήσουμε. δώσουμε το λόγο στους συζητητές. Πρώτα στον κύριο Μπαγιέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως είπατε, είναι πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Είναι φορολογική διαφάνεια το ζητούμενο, θέμα δικαιοσύνη. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε πολυεθνικέ να συγκεντρώνουν ε, κέρδη τα οποία δεν φορολογούνται ενώ οι εργαζόμενοι του, οι ανεξάρτητοι, οι υπεργολαβίε του ε, την κάνουν ε, άλλη και τόσα εκατομμύρια ευρώ διαφεύγουν από το φορολογικό σύστημα των ευρωπαϊκών χωρών. Οπότε, σε αυτό το κείμενο, νομίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει ένα βήμα προόδου, επιτρέποντα να πετύχουμε μεγαλύτερη φορολογική ισότητα. Οι εκθέσει αναχώρα πρέπει να περιλαμβάνουν στοιχεία και για αυτέ τι επιχειρήσει και είναι σημαντικό αυτό για την καταπολέμηση τη προδιαφυγή και φοροαπάτη διεθνώ, αλλά και την ε, ε, υποβάθμιση, την ταχεία υποβάθμιση των ευρωπαϊκών φορολογικών συστημάτων. Να υπογραμμίσω ότι κοιτάζουμε και τον μακρινότερο ορίζοντα με την οδηγία αυτή, με ένα σύστημα προλογικό που να καλύπτει τα στοιχεία τα εθνικά και τα διεθνή. Να υπάρχει μια ε, κοινή φορολογική διακυβέρνηση μεταξύ των χωρών και κοινέ ε, ευθύνε κοινωνική διάσταση των πολυεθνικών εταιριών. Με την συνάδελφο Εύλιν Ρέγνερ έχουμε φιλόδοξε φιλόδοξες για να αλλάξει το ευρωπαϊκό σύστημα με, τρεις, ε, με τρία βασικά στοιχεία. Πρώτον, κυρίω να κοιτάξουμε μια ομάδα πολυεθνικών ε, για να δούμε τα φορολογικά του προνόμια μετά από εξοναχιστικό έλεγχο. Μιλάμε για εταιρείε που ξεπερνούν τον κύκλο εργασιών 40 εκατομμυρίων ετησίω, όπω ε, ορίζουν οι λογιστέ του. 20.000 πολυεθνικές περίπου. 9 στις 10 βέβαια θα εξαιρούνταν αν χρησιμοποιούσαμε άλλο κατόφλι. Γι' αυτό με όσα ανακαλύψαμε ε, φροντίσαμε να χρησιμοποιήσουμε το κατάλληλο κατόφλι. Ε, δεύτερο σημείο, μαύρο μαύρος κατάλογος την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο επίπεδο της Επιτροπής ΕΚΟΝ θέλαμε να υπάρχουν αυστηρά κριτήρια για τον κατάρτιση ενός τέτοιου καταλόγου, αλλά στην έκθεση αυτή θεωρούμε ότι είναι σκοπιμότερο οι πολυεθνικέ να παρέχουν τι δραστηριότητε του σε κάθε δικοδοσία ξεχωριστά εφόσον έχουν λειτουργία σε αυτή ε, και εντό και εκτό Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο μακριά από την πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι Θέλουμε να καλύψουμε διεθνώ την δραστηριότητα των πολυεθνικών και των φυλατρικών του. Θέλουμε να λειτουργήσει καλύτερα η ενιαία αγορά κατά αυτόν τον τρόπο. Και τέλο, στο κείμενο προτείνουμε, ξαναείδαμε τα δεδομένα που προτείνουν οι πολυεθνικέ από μόνε του, με στόχο να υπάρξει φορολογική ενοποίηση και αποτελεσματικά οι χώρε να λαμβάνουν το φορολογικό εισόδημα που του αναλογεί, διευκολύνοντα και απλουστεύοντα και τι ε, διοικητικέ διαδικασίε. Το κείμενο είναι πολύ σημαντικό. Ελπίζω να ενανθεί το κοινοβούλιο πίσω από τι δικέ μου προτάσει και τη Εύελιν, γιατί οι πολίτε μα περιμένουν, περιμένουν αποτελέσματα σε αυτό το επίπεδο. Ε, Κυρίω μια παρέμβαση δική μα ισχυρή και ε, με πυγμή. Σα ευχαριστώ για το χρόνο, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. <clears throat> Κυρία Ρέκνερ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σύμφωνο πλήρω με τα όσα είπε ο Κυπεγέ οι επιχειρήσεις έχουν και κοινωνική ευθύνη. Έχουμε την αρχή της ε, κοινωνικής οικονομίας της αγοράς που αναφέρεται και στη συνθήκη της Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις βεβαίως στόχο έχουν να βγάζουν κέρδη, είναι σαφές, αλλά πρέπει να εκπληρώνουν και τις ε, υποχρεώσεις τους όσον αφορά τις αναφορές και έχουμε διάφορα πράγματα, είτε μιλάμε για non-financial reporting, είτε για τον εξορρυκτικό τομέα. Και βέβαια η δουλειά που έχει κάνει ο Σέρτζο Κοφεράτη για τους μετόχους. Και εδώ πέρα έχουμε ακριβώς την αρχή της δημόσιας αναφοράς τέτοιων πληροφοριών. Είναι αυτό το οποίο είπε ο Ιγκ, να συμπληρώσω και εγώ το κατόφλι, ένα πρώτο κριτήριο τα 750 εκατομμύρια είναι κατανοητό αυτό το οποίο πρότεινε η Κομισιόν κοιτώντας την BEPS αλλά αν δούμε ακριβώς ε, τις ευρωπαϊκές εταιρείε έχουμε ορίσει κάποια κατόφλια εδώ και κάποια χρόνια και δεν έχει νόημα τώρα να μιλάμε εδώ πέρα για 750 εκατομμύρια και θα πρέπει να ανταποκρίνονται και στα υπόλοιπα νομοθετικά κριτήρια. Το άλλο το οποίο προτείναμε βεβαίως είναι οι πληροφορίες οι οποίες θα δίδονται και αφορούν και την γεωγραφική έδρα, τον αριθμό των υπαλλήλων και θα πρέπει να διευκρινιστούν όλα αυτά. Νομίζω είναι κάτι το απολύτως απαραίτητο αν σκεφτούμε και τον στόχο αυτής της έκθεσης και τελικά θεωρώ εγώ η σημαντικότερη απέτηση όταν μιλάμε για τα συγκεντρωτικά δεδομένα. Στόχος είναι ότι οι επιχειρήσεις όπως πρότεινε η Κομισιόν πρακτικά να, ότι έχουν να δίνουν αυτές τις προφορίες μόνο εντός της Ένωσης. Είναι κάτι το οποίο προκαλεί στρέβλωση. Ε, δεδομένου ειδικά του περιβάλλοντος στο οποίο κινόμαστε με την κυβέρνηση Τραμπ και όσο συμβαίνουν και στον υπόλοιπο κόσμο είναι απολύτως απαραίτητο να έχουμε αυτές τις πληροφορίες για την κάθε χώρα. Και χοντρικά νομίζω ότι η ουσία των ε, πληροφοριών αυτών ε, νομίζω θα είναι ακριβώς και το τι γίνεται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένουμε βέβαια πληροφορίες και την συνεργασία με τους συναδέλφους. Ευχαριστώ Εύελιν. Νομίζω μπορούμε να περάσουμε στους σκιώδεις τον κύριο Ροζέτη. Ναι, κύριος Μπάλτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματος του κυρίου Ροζάτη θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους δύο συνζήτες και να σημειώσω το, κάποια πράγματα στο σχέδιο έκθεσης. Μου είπε λοιπόν να παρουσιάσω τα εξής ο κύριος Ροζάτη. Θεωρούμε λοιπόν εδώ πέρα πως δέκα μήνες μετά την πρόταση της ε, Κομισιόν Έχουμε το πρώτο σχέδιο έκθεσης ε, και υπογραμμίζουμε πως η διεθνής ατμόσφαιρα πλέον διαφέρει σε σχέση με όταν δημοσιεύτηκε η πρόταση αλλά εμείς ως ΕΛΚ θέλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτά τα οποία ζητάει το κοινό για να καταπολεμήσουμε την φόρο διαφυγή, την φόρο αποφυγή και τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών εταιριών και το επενδυτικό κλίμα. Ξέρουμε βεβαίως πως η μάχη αυτή δεν μπορεί να την δώσουν μόνα τους ε, τα κράτη-μέλη αλλά ούτε και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό είμαστε υπέρ της ε, διεθνούς ε, συνεργασίας για τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό υπό την αιγίδα του BEPS του ΩΣΑ και μία από τις δράσεις ε, της BEPS είναι η δράση 13 που αφορά τις εκθέσεις αναχώρα η οποία βεβαίως ε, υπάρχει και στην ε, σχετική οδηγία 4 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρέπει να πω ότι εμείς στο ΕΛΚ θεωρούμε ότι ακριβώς η δουλειά του ΩΣΑ πρέπει να αποτελεί τη βάση για την περτέρω δική μας δουλειά για φορολογική διαφάνεια. Θα ήθελα λοιπόν να αναφέρω μόνο κάποια πράγματα που δυσκολεύουν το ΕΛΚ. Όπως ξέρετε, η πρόταση της Κομισιόν έχει ένα κατόφλι 750 εκατομμυρίων τζίρου για να θεωρηθεί μια εταιρεία μεγάλη ή ένας μεγάλος όμιλος ο οποίος θα πρέπει να δημοσιεύει εκθέσεις αναχώρα. Και αυτό είναι και το κατόφλι που προτείνει ο και καθώς ο ΣΑ βεβαίως ε, επιχειρηματολογεί με βάση αυτό το όριο θεωρεί ότι έτσι θα καλυφθεί περίπου το 90% του τζίρου των επιχειρήσεων. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν θα επηρεαστούν και κατά τη διάρκεια των ψηφοφοριών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιμείναμε σε αυτό το κατόφλι, δεν θέλαμε να το κατεβάσουμε έτσι ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που λειτουργούν διασυνοριακά να μην επηρεάζονται. Έχουμε βεβαίως ε, τώρα την πρόταση των συνσηγητών, το να το κατεβάσουμε όμως θα δημιουργήσει όλο ένα παραθυράκι στο σύστημα. Και επειδή εγώ είμαι και σε αυτήν την επιτροπή και στην επιτροπή ε, που αφορά την, τον Πάναμα, ε, βλέπουμε ότι τα παραθυράκια και οι ασυνέπειες είναι αυτά τα οποία δημιουργούν τα κενά τα οποία εκμεταλλεύονται αυτοί οι οποίοι θέλουν να αποφύγουν τους φόρους. Βλέπουμε λοιπόν πως θα πρέπει να ανταποκριθούμε στις απαιτήσει του κοινού χωρίς να βλάψουμε την ανταγωνιστικότητα των εταιριών και άρα θα πρέπει να εστιάσουμε πολύ περισσότερο στην τέταρτη οδηγία και άρα οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να ανταλλάσσονται μεταξύ των φορολογικών αρχών των κρατών μελών. Και βεβαίω το ενδιαφέρον είναι ότι είχαμε και περαιτέρω πληροφορίες που θα γίνονταν δημόσιες. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει το κοινό περισσότερες πληροφορίες από τις φορολογικές αρχές λαμβάνοντα υπόψη βεβαίω τι πιθανέ αρνητικέ συνέπειε για την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών εταιριών και τι περαιτέρω επενδύσει στην Ένωση, το ΕΛΚΑ έχει σοβαρέ επιφυλάξει. Τέλο, ενώ η Κομισιόν θέλει οι πληροφορίε αυτέ να παρουσιάζονται χωριστά ανά κράτο μέλο και για κάθε φορολογική επικράτεια που είναι στην μαύρη λίστα που συντάσσεται, και συνολικά για τις υπόλοιπες ε, φορολογικές ε, επικράτειες, οι συνεισηγητές θέλουν να υπάρχει αυτό ανά αυτό ε, λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο των πληροφοριών πάρα πολύ απλά θα σκότωνε την οποιανδήποτε ανταγωνιστικότητα και την διάθεση επένδυσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι θα πρέπει να έχουμε μια ισορροπημένη πρόταση αποφεύγοντας όμως την υπερβολική τη γραφειοκρατία. Στηρίζουμε λοιπόν την πρόταση των συνεισηγητών για ένα κοινό υπόδειγμα τέτοιων εκθέσεων και αυτό μαζί με την δημοσίευση αυτών των εγγράφων σε κάποια από τις επίσημες γλώσσες θα δημιουργήσει σε λιγότερες παρεξηγήσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση και πάλι θέλει να πρωτοπορήσει σε κάποιο σημείο. Τώρα λοιπόν το θέμα αυτό είναι η φορολογική διαφάνεια. Να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν. Το ΕΛΚ είναι υπέρ της φορολογικής διαφάνειας. Αλλά να είμαστε και ρεαλιστές. Δεν μπορούμε να προετοιμαζόμαστε εμείς για sprint όταν οι άλλοι πηγαίνουν με το πάσο τους. Εδώ απαιτείται διεθνή συνεργασία και όχι μόνο η δική μα φιλοδοξία, η οποία τελικά μπορεί να βλάψει μόνο τις δικές μας εταιρείε και το επιχειρηματικό κλίμα, που είναι η αρχοκοκαλιά της κοινωνικής οικονομία της αγορά. Σας ευχαριστώ. Η κυρία στέρε Σαραγκούτ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είμαι σκιώδη εισηγήτρια από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και πράγματι, όπως προείπε και ο σύντροφο ε, από την Επιτροπή Οικονομικών σκιώδη εισηγητής ε, και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους συνεισηγητές ε, για το έργο τους και έχω να αναφέρω τώρα αρκετές ιδέες. Πρώτα απ' όλα, αν αμφίβολα, το μονοπάτι που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι αυτό της μεγαλύτερης διαφάνειας για τη φορολόγηση των εταιριών, διότι υποχρέωση αποκάλυψη των πληροφοριών, δημοσιοποίηση των πληροφοριών των μεγάλων ομίλων ε, είναι κάτι που προτείνει η Κομισιόν, ε, μας βρίσκει σύμφωνος, πρέπει να γίνει, είναι θετικό. Απλά τώρα πρέπει να συμφωνήσουμε σε ό,τι αφορά το γράμμα της πρότασης ε, της Επιτροπής, γιατί το πνεύμα της μας βρίσκει σύμφωνος. Η ενιαία ευρωστηνή αγορά σημαίνει ότι θα πρέπει οι εταιρείε να πληρώνουν ε, τους φόρους εκεί που ε, δημιουργούν το κέρδος τους και οι πληροφορίες που δίνουν θα πρέπει να οδηγήσει σε περισσότερη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τις φορολογικές πρακτικές. Ταυτόχρονα θα γνωρίζουμε, και αυτό είναι επίσης μια από τις προτεραιότητες της Κομισιόν, Με την υποχρέωση λοιπόν δημοσιοποίηση θα γνωρίζουμε, θα γνωρίζουν οι πολίτε περισσότερο και θα μπορούν να ξέρουν ποια είναι η φορολογική συμπεριφορά των πολυεθνικών. Και έτσι θα αναγκαστούν και αυτέ να πληρώνουν φόρου ε, στη χώρα που ε, δημιουργούν τα κέρδη του. Τώρα, πρέπει να συμφωνήσουμε. Ποιο θα είναι το κατόφλι. Η πρόταση τη Κομισιόν είναι 750 εκατομμύρια. Οι συγκητέ 40 λένε. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει μια τεράστια διαφορά μεταξύ των δύο προτάσεων. Σίγουρα η έκθεση της ε, ΕΟΚΕ λέει ότι είναι μάλλον υψηλό το κατόφλι των 750. Ε, το 40 ε, πρέπει να δούμε και ότι είναι το 9% το όγκου του κύκλου εργασιών. Μεταξύ των δύο κάπου πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία. Επίσης είναι αλήθεια ότι η πρόταση της Κομισιόν δεν επιβάλλει νέο φόρτο στι μικρομεσαίες επιχειρήσει και σέβεται και το επαγγελματικό απόρριτο. Δεν θα πρέπει να χάσουμε σε ανταγωνιστικότητα, το είπε και ο σύντροφο πριν. Και πρέπει να διατηρηθεί η εμπιστευτικότητα, ούτε πρέπει να αυξηθεί το διοικητικό άχθο. Η πρόταση των εισηγητών διαφοροποιείται από αυτήν τη Κομισιόν και σε ένα άλλο σημείο. Εκεί που μιλάμε για τι δηλώσει. Δηλαδή, η πρόταση της Κομισιόν μιλά για την ανάγκη δημοσιοποίηση των εκθέσεων αναχώρα από κάθε φορολογική δικαιοδοσία, ε, όπου δηλαδή και αν δραστηριοποιούνται έστω και εκτό τη Ένωση. Αυτό δεν το λένε οι εισηγητέ. Αλλά η Κομισιόν στρέφεται και στου φορολογικού παραδείσου και σε άλλε χώρε. Και αυτό είναι μια διαφοροποίηση σε σχέση με την πρόταση των εισηγητών που θα πρέπει να δούμε πώ θα αντιμετωπίσουμε. επίση ό,τι αφορά την νομική βάση, στο Συμβούλιο υπάρχει μια διαφοροποίηση αν θα είναι το 50 ή το 115 ε, άρθρο τη συνθήκη η νομική βάση. δηλαδή κανονική ή ειδική διαδικασία. Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε και αυτό. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θεωρώ ότι είναι λογική. Νομίζω ότι είναι αφετήρια διαπραγμάτευσης. Οι εισηγητές και οι σκιώδει νομίζω θα μπορέσουμε να συνεννοηθούμε και να μειώσουμε τις μεταξύ μα διαφορές. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε. Και τώρα από τους συνδετικούς και μεταρρυθμιστές Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Συνολικά η έκθεση είναι καλογραμμένη και καλύπτει τις σημαντικότερες πτυχές της πρότασης της Κομισιόν. Το σοβαρότερο πρόβλημα είναι ότι η Κομισιόν θέλει να περιορίσει τις αναφορές μόνο σε εταιρείε με καθαρό τζίρο που ξεπερνά τα 750 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ η έκθεση είναι πολύ σωστή όταν συνδέει το ε, υποχρέωση αναφοράς ε, με τον ορισμό μεγάλης εταιρείας που υπάρχει ήδη στην περιφερειακή οδηγία. Θα ήθελα να αφαιρθώ λοιπόν στην τροπολογία 6, όπου λέει ότι θα πρέπει τα συνδικάτα και οι υπάλληλοι πολυεθνικών εταιριών να ενημερώνονται για τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται σε ε, βάση πλήρους ε, εργασίας, ε, τα κέρδη της εταιρείας και τον φόρο εισοδήματος. Επίσης οι τροπολογίες 16 έως 30 προτείνουν πάρα πολύ σημαντικές επεκτάσεις σε αυτά τα σημεία, όμως μπορούμε να αναρωτηθούμε τι σημαίνει η τροπολογία 24 που μιλάει για δημόσιες επιδοτήσεις και αν είναι αρκετά ε, λεπτομέρειες. Μήπω θα έπρεπε να λέει δημόσιες επιδοτήσεις και φορολογικές εκτόσει μεταξύ των οποίων και το ύψος και η διάρκεια τους ή κάτι τέτοιο. Τρίτον, θα ήθελα να αλλάξουμε κάποια εκτιμώντας. Στην τροπολογία BEPS ε, του ΩΣΑ ε, που αναφέρουμε θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι δεν έχει επιτύχει τους στόχους της επιπλέον. Το εκτιμώντας 5 μιλάμε για εταιρική ευθύνη. Όπως θα πρέπει να μιλάμε για εταιρική λογοδοσία και αντί για δικαιότερο φορολογικό ανταγωνισμό να λέμε να μην υπάρχει εκμετάλλευση των φορολογικών συστημάτων. Τέλος είναι καλό το ότι αναφέρεται τα ανοιχτά δεδομένα. Θα έπρεπε ίσως να αναφέρουμε το ότι τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να μπορούν να διαβάζονται και από υπολογιστέ. Λοιπόν, να πω επίση πω αυτή είναι η δική μου άποψη και ίσω να μην α, καλύπτει την άποψη όλων των μελών του ECR. Ο κύριος Καλμπέ Σαμπόν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Συμπρόεδρε. Πρόκειται για την αφετηρία, ελπίζω βέβαια να πάμε πιο γρήγορα. Είναι εξαιρετική αφετηρία βέβαια και όλη η δουλειά που έγινε μέχρι τώρα. Το θέμα είναι όμως που πρέπει να εμβαθύνουμε. Εκεί υπάρχουν ε, κάποια ερωτηματικά. Εγώ θα επιμείνω σε αυτά που θεωρώ ότι βρίσκουν σύμφωνους όλους τους παρόντες. Ότι δηλαδή στόχος μας είναι η αύξηση της διαφάνειας και εφαρμογή, ιδέως εφαρμογή του ΜΠΕΠΣ όπως το λέμε και της διαφάνειας και της δικαιοσύνης. Σε ό,τι αφορά τη φορολογική δημοσιονομική ικανότητα και ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν πιο εύκολα να φοροαποφύγουν, για να μην μπορούν να φοροδιαφύγουν. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει απλά να βρούμε τον πλέον πρακτικό τρόπο και το πιο επίγοντα και αποτελεσματικό τρόπο. Με αυτήν την έννοια προτάσεις που διατυπώνουν οι συγητές, πρέπει να πω βέβαια ότι προηγήθηκε ένα έργο, ένα συγγνώμη έγγραφο του Κοινοβουλίου για τον Μπέρπς που και εκεί μου και εισηγητής και ακολουθεί αυτό το ε, κείμενο τώρα. Υπάρχει δηλαδή ένα έδος προηγούμενου και νομίζω ότι μπορούμε να πάμε και πιο πέρα ε, σε σχέση με αυτά που είπε ο ΣΑ. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι και τα πράγματα πηγαίνουν ε, γρήγορα. Είχαμε την Επιτροπή Πάνα, ήρθε ο κύριος Τραμπ και πολλά άλλα έχουν συμβεί. Για όλους αυτούς τους λόγους πρέπει να είμαστε θα έλεγα ρηξικέλευθη στην Ευρώπη, αλλά ταυτόχρονα και ευφύης. Θα αναλύσουμε λοιπόν τώρα ποια είναι τα επίμαχα σημεία μαζί με τους άλλους συντρόφους. Και θα δούμε πού μπορούμε να βρούμε κάποια σημεία ισορροπία για να είμαστε αποτελεσματικοί και να μην βλάψουμε την αναγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Πέντε σημεία βλέπω εγώ για τα οποία θα πρέπει να γίνει κάποια συζήτηση. Ο υποφαινόμενος ε, τουλάχιστον, αλλά και η ομάδα Άλντε. Ε, λοιπόν, ε, θεωρεί ότι πρώτον για τα 750 εκατομμύρια λένε 40 εκατομμύρια. Εγώ θα ζητούσα αυτοί που λένε τα 40 εκατομμύρια να μα εξηγήσουν γιατί επέλεξαν αυτόν το αριθμό. Τι πλεονέκτημα μπορεί να έχει το να μην έχουμε αυτή την πολυεθνική αναφορά ε, των 750 εκατομμύρων που είναι αναφορά από τον ΩΣΑ. Μπορούμε να μην το επιλέξουμε, αλλά γιατί 40 και όχι 60 και όχι 100, αυτό θέλω να μου πείτε επίσης από συγκριτικής πλευράς. Πόσες παραπάνω πολυεθνικές θα περιλαμβάνει αν αυτό το ε, αξίζει ε, ή θα είναι περιφερειακό μόνο το αποτέλεσμα. Δεν είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση προς το παρόν, απλά νομίζω ότι θα πρέπει από τεχνικής πλευράς να δούμε την πλέον ευφυή πρόταση. Επίσης, ο κατάλογος που προτείνεται στο εξαιρετικό έγγραφο των συνεισυχητών μας. Μήπως είναι πάρα πολύ υπερβολική και δυσκίνητη. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη για να ξέρουμε αν μιλάμε για μια εικονική εταιρεία, για κάτι άλλο σοβαρό. Δηλωθέν κεφάλαιο δηλαδή αριθμό υπαλλήλων που απασχολείται σε μερική και σε πλήρη απασχόληση και υλικά ε, περιουσιακά στοιχεία. Μπορεί να είναι υλικό παραγωγής, δεν μιλάμε δηλαδή ε, για τα γραφεία μόνο. Όλα αυτά είναι σημαντικά και ήδη βλέπουμε πολλά πράγματα. Βέβαια το τέλειο είναι εχθρό του καλού και νομίζω ότι ε, δυσκίνητος θα γίνει ο έλεγχος με το να προσθέσουμε και πολλά άλλα στοιχεία. Αυτά νομίζω αρκούν. Αυτό το ε, ενιαίο υπόδειγμα, το, το τυποποιημένο έντυπο, θεωρούμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό να μην παρουσιάζει ο καθένας με το δικό του στυλ και όπως θέλει και ό,τι θέλει, γιατί έτσι ανοίγουμε άλλο ένα παράθυρο και άλλη μία πόρτα ε, στα πολύ καλοπληρωμένα γραφεία των ε, πολυεθνικών για να βρουν λύσεις. Είναι καλή η ιδέα λοιπόν αυτό το υποποιημένο έντυπο. Θέλω, δεν αποφαίνομαι, απλά θέλω να τονίσω αυτά τα σημεία. Βέβαια, εκεί που λέμε ότι είμαστε σύμφωνοι, είμαστε με το αυτό το έντυπο, το υπόδειγμα το ενίο. Αλλά κάτι άλλο στο οποίο πρέπει να εμβαθύνουμε και επειδή θίγεται και η αξιοπιστία της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, ρωτώ, τι νόημα έχει να μιλάμε για ομαδοποιημένα στοιχεία όταν μιλάμε για τον υπόλοιπο κόσμο, εκτός από σφαλικούς φορολογικούς παραδείσους, γιατί νομίζω ότι χάνονται πάρα πολλές πληροφορίες. Και δεν ξέρω και αν είναι και αχρίαστο και αν δεν προκαλεί και σύγχυση. Να έχουμε ένα δεύτερο γύρο ερωτήσεων για το πώς, το πού και τι και πώς. Δεν ξέρω γιατί το επιλέγει αυτό η Κομισιόν. Θα έχει τους λόγους της φαντάζομαι και θα ήταν καλό να ακούσουμε τι έχει να μας πει. Επίσης θεωρώ ουσιαστικά ότι θα πρέπει να καλύψουμε όλο τον κόσμο ουσιαστικά, διότι αν αρχίσουμε να δημιουργούμε κάποια τμήματα όπου υπάρχει αυτή η δήλωση, αυτές οι εκθέσει και κάποια που δεν υπάρχει, δεν νομίζω ότι διευκολύνουν τα πράγματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Καλβέ Σαμπόν. Ε, νομίζω ότι πήρα για τον χρόνο του κυρίου Καβαντά. Πολύ ωραία. Περνάμε στην Γκουε. Κανείς EFTD, ούτε. Α, η πράσινη. Με συγχωρείτε. Ο κύριος Ουρτασούν ο κύριος, ή ο κύριος Ντυρό. Θα ξεκινήσει ο κύριος Ουρτασούν για να συνεχίσει ο κύριος Ντουράν. Πολύ σύντομα αυτά πει ο Πασκάλ. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι όλοι πρέπει να έχουμε επίγνωση και νομίζω έχουμε ότι στόχος μας είναι να προωθήσουμε ένα πολύ σημαντικό φάκελο. Και υπάρχουν αυτά τα φορολογικά σκάνδαλα των τελευταίων ετών που μας υποχρεώνουν να είμαστε φιλόδοξοι. Το λέω γιατί η μη νομοθεσία ε, θα μπορούσε να είναι ε, ίσως λιγότερο κακό από το να μην έχουμε την κατάλληλη νομοθεσία, την αποτελεσματική νομοθεσία. Τουλάχιστον αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Έχουμε μια φιλόδοξη πρόταση. Ξέρουμε και τις δυσκολίες που θα έχουμε στο Συμβούλιο, τα είπαμε και πιο πριν, η πρόταση να αλλάξει και η νομική βάση ε, ε, και αυτά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Εγώ θα εστιάσω σε βασικά σημεία. Πρώτον, από τα 750 εκατομμύρια ε, να κατεβούμε στα 40 όσο αυτό το τζίρο, αυτό είναι ένα ουσιώδες θέμα αν θέλουμε να είμαστε φιλόδοξοι. Εμείς θα στηρίξουμε την πρόταση των εισηγητών. Θέλω να του ευχαριστήσω και του δύο για το έργο του. Διότι αν πάμε, ε, όπως είπε και ο με 750, ένα στι 10 πολιτικέ θα μείνουν εκτό. ρύθμιση. Τι νόημα έχει δηλαδή τελικά να έχουμε αυτή τη ρύθμιση, αν είναι για ένα τόσο μικρό αριθμό εταιριών μόνο να ισχύει. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, ή μάλλον δύο σημαντικά άλλα ακόμη στήματα στα οποία θέλω να εστιάσω. Το πρώτο είναι το εξή. Η πρόταση ακομη στηματα στο οποια Κομισιόν, το είπε τη κομισιον το ειπε νομιζω και ο κύριο ε, Καλβέτ, θεσπίζει ότι τα στοιχεία εκτός ένωσης θα είναι ομαδοποιημένα. Εμείς δεν συμφωνούμε. Πρέπει να μην είναι ομαδοποιημένα αυτά τα στοιχεία. Μιλάμε για μια εξοδαφικότητα. Αν δεν έχουμε απομαδοποιημένα στοιχεία, δεν θα μπορούμε να δούμε τι δράση κάνουν στις διάφορες φορικές δικαιοδοσίες οι διάφορες εταιρείε. Τρίτον, στην πρόταση της Κομισιόν υπάρχει ένα παραθυράκι διαφυγής για κάποιες επιχειρήσεις, γιατί λέει ότι σε αν, αν σε κάποιες φορολογικέ δικαιοδοσίε απαιτείται έκθεση αναχώρα εκτός ένωσης, αυτό δεν θα πρέπει να γίνεται στην Ευρώπη. Αυτό πρέπει να αλλάξει, νομίζω. Ως κοινοβούλιο πρέπει να αλλάξουμε αυτό το θέμα, γιατί έτσι δεν θα μπορούν... Ε, να αποφεύγουν τη δήλωση πολλές εταιρείε. Και στηρίζω την πρόταση των ε, δύο συνεισηγητών, επαναλαμβάνω, και όταν μιλάμε για την απώλεια ανταγωνιστικότητα δυνητικά, εμεί λέμε από τι εταιρείε να κάνουν αυτά που ζητάμε ήδη να κάνουν οι τράπεζε. Άρα δεν υπάρχει καμιά απώλεια ανταγωνιστικότητα κατά την άποψή μου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια έκθεση αρκετά σκληρή για έναν οικολόγο. Εμείς που μας αρέσουν οι επικρίσεις, για μια φορά πρέπει να πω ότι είμαστε σε πλήρη συμφωνία και με την έκθεση αυτή και με τη δουλειά των δύο συναδέλφων Μπαγιέτ και Ρέγνερ. Πολύ σοβαρότερα τώρα. Γιατί 40 εκατομμύρια τέθηκε και προηγουμένω το ερώτημα, γιατί απλούστατα είναι ο ορισμό των μεγάλων επιχειρήσεων από την οδηγία περιλογιστικών. Υπάρχει συγκεκριμένο σκοπό λοιπόν και εμείς θα εκφράσουμε ακριβώς την ίδια απέτηση. Όπως πολύ σωστά εξήγησαν οι συνάδελφοι. Πρέπει η ανάγκη διαφάνειας να ισχύσει μόνο για τις μεγάλες επιχειρήσεις και όχι στις ιδιαίτερα μεγάλες. Για όσα υπόθηκαν ε, ως προς την ανάλυση των στοιχείων και τα οποία συμμερίζομαι και μάλιστα έντονα να Επιμένω σε δύο σημεία παρόλο που αναφέρθηκαν γρήγορα. Πρώτον, ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με λογιστική διαφάνεια. Σε καμία περίπτωση δεν ασχολούμαστε με τη φορολογική βάση, τα επιτόκια, του συντελεστέ μάλλον ή οτιδήποτε άλλο. Όχι, στα πλαίσια τη διαφάνεια για του μετόχου θέλουμε να το δούμε. Προκαλεί συζητήσει το θέμα και γι' αυτό είναι και σημαντικό. Είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο να παραμένει σαφέ. Και τελευταίο στοιχείο δεν είναι επικριτικό σχόλιο, μάλλον είναι περισσότερο έκλεισε για προστίκη. Δεν λέγεται τίποτα για κυρώσει, ενδεχόμενε κυρώσει. Αν δούμε στη Γαλλία, πόσο δύσκολο κάποιε φορέ είναι να, αποκτήσει, να πάρει κανεί πληροφορίε. Επειδή δεν υπάρχει καμία αναφορά σε σαφεί κυρώσει σε περίπτωση μη σεβασμού ε, αποστολή πληροφοριών, θα ήθελα και αυτό το σημείο κάπω να καλυφθεί. Πρόεδρο, ευχαριστούμε κύριε Ντυρό. Δεν βλέπω άλλη σκιώδες να ζητούν το λόγο, οπότε να περάσουμε στο ΚΑΤΣΤΙΑΙ. Ο κύριος Φέρπερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν νομικός δεν είμαι. Ένα μέλος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων και ελπίζω να μάθω κάτι από την σοφία των συναδέλφων, αλλά διαβάζοντας την έκθεση δεν ε, έγινα σοφότερος. Έχουμε ε, μεταφέρει την ε, πρωτοβουλία BEPS εμείς ως φορολογικό θέμα. Και εκεί πέρα βεβαίως υπάρχει η έκθεση αναχώρα, η οποία όμως δεν είναι δημόσια και αναρωτιέμαι τώρα πώς θα γίνει νομικός κάτι τέτοιο σε επιχειρήσεις οι οποίες εντάξει μπορεί να είναι πάνω από το κατόφλι των 40 εκατομμυρίων Ε, παραδείγματο χάρη ε, δεν είναι ΑΕ. Εταιρείε ε, όπου οι ιδιοκτήτε είναι μια οικογένεια και ένα άτομο ή δεν είναι εισηγμένο. και θα ήθελα οι νομικοί να με ενημερώσουν. Το δεύτερο. Αυτό είναι θέμα φορολογικό ή εσωτερικής αγοράς. Αν είναι θέμα εσωτερικής αγοράς τότε γιατί ασχολούμαστε με θέματα τα οποία είναι εκτός ε, της ε, εσωτερικής αγοράς και με επικράτειες εκτός της εσωτερικής αγοράς. Πρέπει να δοθούν κάποιες σοβαρές απαντήσεις και βέβαια έχουμε και την μητέρα όλων των ερωτήσεων. Τι θέλουμε να επιτύχουμε. Θέλουμε να απολογηθούν ε, και να στριμώξουμε τις πολυεθνικές μας επιχειρήσεις ή θέλουμε περισσότερη φορολογική ειλικρίνεια γιατί ήμουν εγώ και στην τάξη 1, 2 και στην Επιτροπή του Παναμά, είμαι τώρα, και με το θέμα των πολυεθνικών έχουμε το πρόβλημα του ότι δεν είναι ότι έχουν ιδιωτικούς λογαριασμούς στον Παναμά, αλλά ότι έχουν συνεννοήσεις με κράτη για να πληρώνουν λιγότερους φόρους. Και ο στόχος ε, θα πρέπει να είναι ακριβώς να δούμε ε, ποιος είναι ο τζίρος ε, και οι φόροι που πληρώνονται σε μια χώρα και μετά να έχουμε άρα ένα εργαλείο για να δούμε αν το φόρος πληρώνεται είναι δίκαιο σε σχέση με το τζίρο σε μια χώρα. Αυτός είναι ένας δείκτης, αλλά το θέμα εδώ πέρα ποιο είναι, να αποτρέψουμε άλλες χώρες να κάνουν ειδικέ τέτοιες φορολογικές ε, συνεννοήσεις πρέπει να δούμε και τι γίνεται και με την ανταλλαγή πληροφοριών. Και αναρωτιέμαι λοιπόν αν απαντάει σε αυτό το ερώτημα η έκθεση, μήπως τελικά βάζουμε τρικλοποδιά στον εαυτό μας και εξασθενούμε τελικά τα κράτη-μέλη και κατηγορούμε όλες τις εταιρείε ως δυνητικά ε, φοροφυγάδες, ενώ δεν είναι οι εταιρείε είναι τα κράτη-μέλη ή τα κράτη γενικώ που ευνοούν τις εταιρείε. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μεταξύ μας αυτά τα ερωτήματα πριν αρχίσουμε να μιλάμε για κατόφλια και τέτοια πράγματα. Σας ευχαριστώ κύριε Φέρμπερ. Περβάνος Περές. Σας ευχαριστώ. Να συγχαρώ τους συνεισηγητές γιατί μας δίνουν μια πολύ καλή βάση για τις συζητήσει μας για μια από τις πρόσφατες πρωτοβουλίε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι ουσιώδους σημασίας για μας. Μια μικρή παράκαμψη όμως για να δούμε το ιστορικό της όλης ε, ιδέας και να θυμηθούμε τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησε το Ηνωμένο Βασίλειο για να μην προχωρήσει στα φορολογικά μαζί με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιοι εδώ θα το θυμούνται. Με τις συμφωνίες της ΦΕΙΡΑ Μιλήσαμε για την διαφάνεια στις, στους λογαριασμούς αποταμίευσης ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο είχε πάρει μια ρήτρα εξαίρεση σε αυτό το θέμα όταν υπάρχουν ε, συμφωνίες με τρίτες χώρες. Και είχαμε ξεκινήσει συζητήσεις τότε με πολλούς εξωτερικούς συνεργάτε. Και τώρα περάσαμε σε μια τέτοια διάρθρωση και σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο που αναγκαζόμαστε να ξαναδούμε τα φορολογικά σε ένα άλλο πλαίσιο. Η ίδια αυτή η χώρα, το ΕΒ, Βασίλειο, μας εξηγεί ότι σε κάθε περίπτωση ότι θα κάνει ό,τι θέλει στα φορολογικά. Γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούμε να προχωρήσουμε όλοι μαζί και ω Οικονομική Ένωση. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε φορολογικά μέτρα στο ΕΒ, Βασίλειο, αφόσον εμεί μεταξύ μα καλά-καλά δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ποια είναι, η, ποια είναι τα ρητορικά τέχνα, τεχνάσματα που χρησιμοποιούνται και αξιοποιούνται και σε θέματα φορολογικά και οικονομικά. Αλλά πρέπει λιγάκι να κάνουμε και εμείς τη δική μας προσπάθεια. Ε, πρέπει να κοιτάξουμε να παρακολουθήσουμε πώς αντιλαμβάνονται και οι συμπολίτες μας τα θέματα αυτά του θέματος ας πούμε της αναέκθεσης αναχώρας έκθεσης. Οι πολίτες θεωρούν αδιαφανή αυτό τον μηχανισμό και βλέπουν ότι οι εταιρείε δεν ε, ε, καταβάλουν το ανάλογο φορολογικό τίμημα εκεί όπου παίρνουν τις πρώτες την ε, ουσία της παραγωγής τους ή εκεί που έχουν καταστήσει την έδρα τους δεν υπάρχει καμία αναλογικότητα ενώ αντιστρόφως άλλες εταιρείε κινητοποιούν πολιτικούς ηθήνοντες για να συνεχιστεί αυτό το κρυφτούλι που έχουν ε, διοργανώσει. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να αναφερθώ και σε μια απόφαση που ελήφθη από μια χώρα που γνωρίζω αρκετά καλά, η οποία ονομάζεται Γαλλία, και από το Συνταγματικό Συμβούλιο πρόσφατα, την έχω ακόμα στη μνήμη μου, ελήφθη η απόφαση που λέει ότι η Γαλλία αρνήθηκε να δώσει κάποια στοιχεία στην ε, αναχώρα έκθεση. Όμως, ακριβώς το Συνταγματικό Συμβούλιο ε, της Γαλλίας αναγνώρισε ότι ο στόχος της διαφάνειας και της αναχώρας γνώσης του τι κέρδους έχουν οι εταιρείε έχει συνταγματική διάσταση. Αυτό υποχρεώνει κάθε κατός μέλος έχω την εντύπωση, να προχωρήσει θέλει δεν θέλει και να προχωρήσουμε όλοι μαζί έχοντας υποδειγματική στάση στις διαπραγματεύσεις μας με τα υπόλοιπα κράτη. Ε, ε Ω προ τα βήματα ε, εξέλιξη και πρόοδου που προτείνουν οι συγκεκριτέ, θέλω να σταθώ σε δύο σημεία. Το πρώτο έχει να κάνει με την αλλαγή του ε, ε, ορίου, του κατοφλίου. Είναι πραγματικά, νομίζω, εκπληκτικό ότι ε, χρησιμοποίησαμε έναν αριθμό οδηγιών και πρέπει να βασιστούμε στο αληθοφανές άλλων ε, τομέων για τα 40 εκατομμύρια ας πούμε και το κατά πόσον οι 9 στις 10 πολυεθνικές τη γλιτώνουν. Νομίζω ότι η πληροφόρηση του κοινού είναι σημαντική και ως προς τα ε, λεπτομερή στοιχεία θέλουμε να έχουμε υπόψη ε, και τι αριθμός διαφεύγει από τη φορολογία ως προς τον ε, αρνητικό κατάλογο. Υπήρξαν κάποια πηγενέλα, αλλά νομίζω ότι ο στόχος είναι να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια. Έτσι. Οπότε η προσέγγιση που προτείνεται είναι σωστή. Όσο για το αν το θέμα είναι περισσότερο νομικό ή φορολογικό, νομίζω το θέμα αυτό έχει λήξει. Είχαμε αποφανθεί το φορολογικό είναι η διάσταση που μας αφορά ε, στην αρχή της όλης διαδικασίας, αλλά μετά έχει να κάνει και μετερικό δίκαιο. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το δουν και να το ξεκαθαρίσουν το Συμβούλιο και η Επιτροπή. Ευχαριστούμε, Περβάνης. Ευχαριστούμε. Κάποιος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα αναφερθώ σε δύο μόνο σημεία ουσίας και εν μέρει θα μιλήσω για την νομική βάση. Έγιναν ε, κάποια ερωτήματα και για το πεδίο εφαρμογή και για το κατόφλι της πρότασης που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε ό,τι αφορά την απομαδοποίηση, την ανάλυση των πληροφοριών που θα δημοσιεύονται. Θα εστιάσω στα δύο αυτά σημεία, πολύ σύντομα. Πρώτον, γιατί οθετήσαμε την προσέγγιση αυτή που οθετήσαμε, γιατί ο στόχο ήταν να εστιάσουμε στους πιο προβληματικούς τομείς. Αν δείτε το κατόφλι των 750 εκατομμυρίων εστιάζει σαφώς στις εταιρείες που έχουν και κίνητρο αλλά και την εμπειρία και τα μέσα για επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό. 6.000 περίπου εταιρείε είναι αυτές που υπερβαίνουν το κατόφλι, αυτό τον τζίρο, άρα το 90% των εσόδων που κάνουν οι πλήρες το καλύπτουμε. Εάν κατεβούμε σε αυτό το κατόφλι των 40 εκατομμυρίων με βάση τα στοιχεία των συνεισηγητών αυξάνεται ο ρυθμό των επιχειρήσεων που καλύπτονται τριπλασιάζεται συγκεκριμένο ρυθμός αλλά περιθωριακός θα είναι μόνο ο αντίκτυπος στα έσοδα που θα καλύπτονται από το κείμενο. γιατί μόνο 10% αύξηση ε, της κάλυψης του εισοδήματος είναι δυνατή με βάση τα στοιχεία τόσα. Εμείς λοιπόν επιλέξαμε αυτό το κατόφλι για να είμαστε συνεπείς με την προσέγγιση τη διεθνή, στο πλαίσιο του ΩΣΑ δηλαδή, αλλά και για να είμαστε αναλογικοί στην προσέγγιση μας. Δεύτερο σημείο, την απομαδοποίηση των στοιχείων. Στόχος μας είναι και εδώ να εστιάσουμε εκεί που υπάρχει πρόβλημα στις μη ε, ενωσιακές δικαιοδοσίες, όταν δηλαδή είναι κακή η φορολογική διακυβέρνηση. Και εκεί θα βάλαμε αυτές τις δικαιοδοσίες, θα τις βάζουμε στον κατάλογο. Αν πάμε πιο πέρα, υπάρχει ο κίνδυνος ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να τεθούν ε, σε πάρα πολύ σημαντικό ανταγωνιστικό μειονέκτημα. Γιατί θα πρέπει να δημοσιοποιούν πληροφορίες που οι ανταγωνιστέ τους από τις άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα προβλέπεται να τι δημοσιοποιούν αυτές τι πληροφορίες. Και βέβαια αυτό είναι ζήτημα κόστους αλλά και ζήτημα πληροφόρηση που θα μπορούν να παίρνουν ε, για τις δραστηριότητες των δικών μας επιχειρήσεων οι ανταγωνιστέ μας από μη ευρωπαϊκέ χώρε. Αυτή είναι η γενική προσέγγιση να επανέλθουν συντομία στα κατόφλια. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ότι εστιάζουμε στις επιχειρήσεις με την πρότασή μα που πραγματικά δεν έχουν πρόβλημα, να σας πω ότι όλες οι εταιρείε που αυτή τη στιγμή είναι υπό έρευνα από το τμήμα ανταγωνισμού για πιθανές κρατικέ επιδοτήσει, ε, και φορολογικέ συμφωνίε ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτονται από το κατόφλι που προβλέπουμε στη δική μας πρόταση. Πολύ σύντομα τώρα να επανέλθω στη νομική βάση. Φυσικά και συμφωνούμε απόλυτα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά την νομική βάση. Και ήταν ε, πολύ θετική γνωμοδότηση τη νομική υπηρεσία που ψηφίστηκε στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων τον Ιανουάριο. Και είμαστε απόλυτα σύμφωνοι μαζί σα. Εγώ απλά μια προειδοποίηση. Μην εισαγάγετε τροπολογίε στο κείμενο αν αυτέ δυνητικά θα μπορούσαν να δώσουν στήριξη και επιχειρήματα σε αυτού που υποστηρίζουν ότι δεν έχουμε πλέξει τη σωστή νομική βάση. Φυσικά και επιμένουμε ότι ο στόχο τη πρότασή μα είναι να εξασφαλίσουμε τη διαφάνεια και την λογοδοσία των επιχειρήσεων που καλύπτονται και σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να ε, επηρεάσουμε την εφαρμογή τη νομοθεσία ε, τη Βολή σε εθνικό επίπεδο. Και αναφέρομαι στην αναφορά της εναρμονισμένης προσέγγιση την εφαρμογή των εθνικών φορολογικών συστημάτων δροπολογία τροπολογία 1. Θα έπρεπε να εξετάσουν, νομίζω, από αυτό το πλαίσιο την τροπολογία αυτή οι συνεισήγητες Θέλω πάντως να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές για το έργο τους ε, και σίγουρα προσβλέπουμε στη συνεργασία μας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να προχωρήσουμε στο θέμα αυτό. Έχουμε συνεργαστεί εντατικά και με το Συμβούλιο. Νομίζω είχαμε τουλάχιστον εννέα ε, ομάδες εργασίας ε, με το Συμβούλιο. Έχουμε κάνει και μια τεχνική συνεδρίαση και τώρα θέλουμε να συνεργαστούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να προχωρήσουμε το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι έχουμε πέντε λεπτά για τους συζητητές, αν θέλουν να σχολιάσουν. Έβελιν, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις ε, παρεμβάσεις. Μας διευκολύνουν πολύ στην ε, δουλειά μας. Ε, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την Κομισιόν. Βεβαίως ε, μιλάτε εδώ πέρα να επικεντρωθούμε σε χώρες οι οποίες δεν έχουν επαρκή διακυβέρνηση. Ναι εντάξει αλλά μην δημιουργήσουμε πάλι νέα παραθυράκια. Αυτό ακριβώς θέλουμε να αποφύγουμε. Ειδικά τώρα για τις ερωτήσεις του κυρίου Φέρμπερ και άλλων για τις ε, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Γι' αυτό ακριβώς ορίσαμε το κατόφλι των 40 εκατομμυρίων. Είναι η οδηγία περί αναφοράς, υποχρέωσης αναφοράς, όπου ακριβώς εξαιρούνται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αν δούμε τις οικογενειακές επιχειρήσεις, το θέμα το οποίο θέσατε, βεβαίως όταν είναι τεράστιες επιχειρήσεις και ας είναι και οικογενειακές, αν ξεπερνάνε αυτό το κατόφλι, μιλάμε για την IKEA, δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι μια μικρομεσαία επιχείρηση. Αν ε, ξεπερνάει το κατόφλι πρέπει να καλύπτεται. Παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Δεν, δεν. Δεν έχει διερμηνία. Χουγ. Ευχαριστώ. Ήταν μεγάλη χαρά να φτάσουμε ως εδώ ε, και να έχουμε μπροστά μας τη συνεργασία με τους Κιώδη. Με τα χαρά λοιπόν θα κοιτάξουμε όλα τα θέματα που ε, εντοπίστηκαν. Πολύ ωραία. Φτάνουμε στο τέλος της συζήτησης. Ίσως να πω ότι η προθεσμία για την των απολογιών είναι 15 Μαρτίου. Η εξέτασή τους 3 Μαΐου και η ψηφοφορία στην ΕΚΟΝ σε μεικτή συνεδρία 29 ή 30 Μαΐου. Ευχαριστώ που σεβαστήκατε πλήρως το χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ.